την θαραλέα δήλωση που έκανε η μητέρα του θύματος ε, για την ε, συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ernst Strasser. Εγκατέλειψε ο Ernst Strasser την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 24η Μαρτίου 2011 και σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφια 1 και 3 του κανονισμού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει τη χειρία της έδρασα από την ημερομηνία αυτή. Η κυρία Χέλα Ράνερ εγκατέλειψε την έδρα της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 1η Απριλίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 και παραγράφους 1 και 3 του των κανονισμών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την χειρεύση της έδρασα και από την ίδια ημερομηνία και όλες ε, Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ε, ενημέρωσαν ότι ο κύριος Έρθο Στράσερ αντικαταστάθηκε από τον κύριο Χούμπερτ Πίρκερ από την 31η Μαρτίου 2011. Θέλω να καλωσορίσω το νέο Ευρωβουλευτή και να υπενθυμίσω σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισμού μέχρι ότου θα έχουν ε, επιβεβαιωθεί τα, η, θα έχει επιβεβαιωθεί η εντολή του μέλους και υπό τον όρο ότι θα έχει προσυπογραφεί η γραπτή δήλωση από πλευράς του. Ο κύριος Πίρκερ μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα. Ο κύριος Χούμπερτ Πίρκερ βρίσκεται παρόν στο σώμα. Σας καλωσορίζουμε κύριε Χούμπερτ Πίρκερ. Σας ευχαριστώ. θα θέλατε να παρέμβετε διαδικαστικό από πλευρά σας. Παρακαλώ. Ναι, διαδικαστικό πρόεδρε. Σε σχέση με τον κύριο Στράσερ και τους άλλους που αποχώρησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ίσως ε, υπέστησαν αυτή την κατηγορία ότι ήταν ένοχη διαφθοράς και ότι σε σχέση με τις αποζημιώσεις δεν θα έπρεπε να καταβάλλονται. Όταν κάποιος καταγγέλλεται λόγω διαφθοράς ε, δεν μπορεί να παίρνει τέτοιου είδους επιδόματα. Παρακαλώ να το προσέξετε αυτό. Ε, Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Δεν ήμουν έτοιμος να απαντήσω αυτή την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Ο κύριος Μάσιπ, διαδικαστικό κύριε Μάσιπ, διαδικαστικό πρόεδρε. Εσείς αναφερθήκατε εξ ονόματος όλων των Ευρωβουλευτών ότι σε σχέση με ένα κράτος, το, μια πολιτεία των ΗΕ θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτήν για την ε, αντικατάσταση της θανατικής ποινή ε, με την ποινή των, ε, της ισοβίας φυλάκισης. Εντάξει, αλλά να, όχι σε σχέση με την ε, ε, καταδίκη σε ισόβια όπως ε, υφίσταται στις ΗΠΑ θα πρέπει να πούμε ότι θα μετατραπεί η θανατική ποινή με μια άλλη αναλογική ποινή που θα επιβάλλεται στον καταδικαστέντα σε θάνατο. Σας ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί αφεαυτού ξεχωριστά αυτό τελώς. Δεν είναι δυνατόν έτσι να ληφθεί μια απόφαση αυτό σχέδια.